Αγαπητοί συνάδελφοι, άρχεται η συναντρίαση. Εάν δεν έχετε αντιρρήσει, θεωρείται εγκεκριμένη ημερησία διάταξη. Θυμίζω ότι οι αποφάσεις των συντονιστών της 21ης Φεβρουαρίου ε, βρίσκονται στα, πρακτικά, στα δοσιέ σας και αν δεν έχετε καμία αντίρρηση θεωρούμε ότι επίσης ε, εγκρίνονται οι αποφάσεις των συντονιστών. Θα περάσουμε τώρα μέσω στην ψηφοφορία. Παρακαλώ βάλτε τις κάρτες σας στα μηχανήματα. Για να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Από ό,τι φαίνεται όχι όλοι ακόμα. Η κυρία Τωμά. Έχασα την κάρτα μου. Επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, δεν φέρνουμε κάρτα. Très Καλώς. Πέρασε. Πολύ ωραία πλειοψηφία. Και πολλές άποχες. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Την έκθεση κατευθυντήριες οδηγίες για τον προπολογισμό του 2019 του κυρίου Ντανιέλε Βιώτη, τον οποίο και δεν βλέπω. Πού είστε? Χρόνια σας πολλά, είναι τα γενέθλιά σας σήμερα. Ευχαριστώ. Ελπίζω να μου κάνετε δώρο. Yeah, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ψηφίζουμε συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έχουμε τώρα την τροπολογία υπαριθμών 38 υπέρ ε, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές αυτό. Ας το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρασα. Εγκρίνεται. 18 είπε. Εγκρίνεται, εν πάση περιπτώσει. Ήταν η τροπολογία παριθμών 41 αυτή. Συμβαστική 4. Υπέρ. Υπέρ 4 συμβαστικής. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αυτό θέλει επαλήθευση, παρακαλώ. Να ψηφίσατε όλοι, πέρασε τις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 17-12. Η τροπολογία υπάρχει 53 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά άποχες αυτό θέλει έλεγχο παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει τώρα πέρασε εγκρίνεται 16 υπέρ 13 κατά Ποια ήταν αυτή, η 55. Συμβαστική 5, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 63, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική παρήθμο 8 υπέρ κατά Αποχές δεν κρίνεται. Η τροπολογία 86 π. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έχουμε την τροπολογία 95 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 98 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 134 τώρα. Βλέπετε εδώ τι γίνεται. Σε τέσσερα τμήματα. Και προφορική τροπολογία. Το πρώτο τμήμα. Η προφορική είναι στο τρίτο. Θα ψηφίσουμε όμως με τη σειρά, έτσι. Πρώτο τμήμα, λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το τρίτο, με την προφορική, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και το τέταρτο, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 135, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 136 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 138 το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τρίτο τμήμα ορίστε Τσεκ. Καλά. Θα επαληθεύσουμε το δεύτερο τμήμα, παρακαλώ, τη 138. Αρχίζει η ψηφοφορία τώρα. Πέρασε. Απορρίφτεται. 12 υπέρ, 20 κατά. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το τέταρτο υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στην 142 όμως έχουμε διάφορα τμήματα να ψηφίσουμε εκτός συμβιβασμού. Το τρίτο τμήμα υπέ. κατά, Επαλήθευση παρακαλώ. Ψηφίζουμε στην τροπολογία 142 το τρίτο τμήμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασα. Εγκρίνεται. 17 υπέρ 11 κατά. Και έχουμε και ένα τέταρτο τμήμα υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται αυτό. Τσεκ. Ας το τσεκάρουμε λοιπόν, αρχίζει τώρα η επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται, 17 υπέρ, 11 κατά. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 21 υπέρ κατά εγκρίνεται 22 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβαστική 23 υπέρ κατά εγκρίνεται η τροπολογία 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 152 υπέρ κατά Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά στο ελέγξουμε για καλό και για κακό. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. 17 17-15 εγκρίνεται. Ποια ήταν αυτή, 152, 153 τώρα είπε. Κατά. εποχές εγκρίνεται. 154 είπε. Κατά. εποχές απορρίπτεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Η τροπολογία 1 είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. δύο σε τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία τρία έχει καταπέσει αφού οι δύο εγκρίθηκε. Ναι. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία μόνο 6 υπέρ. Α, όχι, έχει καταπέσει αυτή. 24 συμβιβαστική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του κειμένου τώρα αποστροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση που αρχίζει τώρα. Πέρασα. Εγκρίθηκε 26 ψήφοι υπέρ, 4 κατά και 3 αποχές. Ορίστε, να το δώρο σας για τα γενέθλιά σας κύριε Βιώτη. Συγχαρητήρια. Ωραίο δώρο σας κάναμε mise en œuvre de l'instrument de εφαρμογή του μέσου αναπτυξιακής συνεργασίας ανθρωπιστική βοήθεια Ευρωπαϊκό, Κοινων... Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης Χορδί Σολέ υπαριθμόν 1 υπέρ κατά Αποχές απερίφθη 2 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 7 υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές απεριφθή 9 υπέρ κατά αποχές και θα επαληθεύσουμε αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 9 ψηφίσατε όλοι πέρας απερίφθη 19 κατά 12 υπέρ Υπαριθμόν 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική υπαριθμόν 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές και επαληθεύουμε τη 15 αρχίζει Πέρας. Απέριφθη 19 ψήφοι κατά, 12 ψήφι υπέρ. Υπαριθμών 17 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά Α, κατέπεσε, συγγνώμη, 21 υπέρ. Κατά. Αποχές και επαληθεύουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Και εγκρίνεται 15 ψηφι υπέρ, 14 κατά. Η υπαριθμόν 21 ήταν αυτή. Υπαριθμών 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ. Κατά. Αποχές και για το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε ονομαστικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Και έγκρινατε 26 υπέρ, 3 κατά, 3 αποχές και συγχαρητήρια στο χώρο της Ολέ. κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, έκθεση τη ε, κυρία ε, Κρέσλε. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Τροπολογία 2. Τροπολογία 2 αφορά την παράγραφο 2α9. Ναι. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κύριε Βίλαντ. Πρόεδρε, τουλάχιστον στο γερμανικό κείμενο, στην πρώτη τροπολογία, ε, ακούσαμε τροπολογία υπαριθμών 2 και την υπερψήφισα. Αυτό άκουσα τουλάχιστον τη διερμηνία. Αυτό εννοούσατε. Δύο μου είπαν εμένα πάντως. Τροπολογία 1 είναι στο τέλος του, του καταλόγου ψηφοφοριών αφορά τη λογική σκέψη ε. Η 1. Τροπολογία 2 λοιπόν. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε εγκρίνεται 16-12. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 αποσύρεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 9 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 10 με μια διευκρίνηση τεχνικού ύφου ε, τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 αποσύρεται τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά θα κανω παληθευση επαλήθευση ηλεκτρονική επαλήθευση ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 17-13 τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. το Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. το Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. το Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται για όλο το κείμενο ονομαστική ψηφορία που άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται 28-3. Συγχαρητήρια στην Πρόεδρο Κρέσσα. Vient ensuite... Euh, Μετά έχουμε μεταφορά παρουσιάζει ο συνάδελφος Μουρεσάν, Γενικο Συγητή και είναι συνέπεια της ψηφοφορία Ο κ. Μουρεσάν αποσιάζει, δικαιολογημένα. Η μεταφορά που προτείνεται λαμβάνει υπόψη τα αποτέλεσμα ψηφοφορία για το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση με ηλεκτρονική ψηφοφορία που άρχεται. Ο κ. προτείνει θετική ψήφο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε εγκρίνεται 23 με 4 για τα άλλα τμήματα τώρα έχουμε τροποποίησεις ο Ρίτσοντ Άσουεθ θα μας παρουσιάσει τις συστάσεις του για την τροποποίηση του σοφατά στελέχη μικρή αλλαγή που ζήτησε ο διαμεσολαβητής ε, ένα ST7 μόνιμη και ένα SD, μια θέση SD και έτσι μπορεί άλλος, ε, άλλο ένα μέλος να προσληφθεί για εξέταση υποθέσεων εμπίπτει στο άρθρο 50 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, που τεχνικός δεν χρειάζεται ψηφοφορία. Παρόλο που συστήνω έγκριση, σημειώνουμε λοιπόν ότι η μεταφορά που προτάθηκε ε, εγκρίνεται την προτείνουμε να εγκριθεί. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά, Ρίτσαρτ Άσφουεφ. Σκιώδηση εισηγητές έχουν κάποια παρατήρηση, δεν βλέπω αν υπάρχει παρατήρηση. Συνεπώς, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα θεωρηθεί ότι αυτή η πρόταση συγκρίνεται. Στρέφομαι προς την Μόνικα Χολμάιερ. Δεν ζητήσω για την πολιτική για τα ακίνητα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν. την ψηφοφορία, τις ψηφοφορίες μας μάλλον. Μόνικα, δεν έχετε κάποιες πληροφορίες που θα θέλατε να κοινοποιήσετε στην Επιτροπή. Όχι. Την επόμενη φορά. Ωραία. Τώρα έχουμε τα πιλωτικά προγράμματα και προσκευαστικές δράσεις. Προϋπολογισμός 2018 και τον επόμενο προπολογισμό του 2019. Και ο Σμουρεσάν απουσιάζει. Ο Ντανιέλ Εβιώτη θα μας μιλήσει καταρχάς για 2019. Και έτσι θα θυμηθούμε και τι συνέβη το 2018. Κύριε Γενικέ εισηγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βεβαίως δεν έχουμε πολλά να πούμε ακόμα για τα πιλωτικά σχέδια για το 2021. Απέχουν ακόμη πολύ από την περίοδο, απέχουμε ακόμα πολύ από την περίοδο παρουσίασης συζήτησης ε, των προτάσεων της Επιτροπής ε, και δικών μας συμπερασμάτων, αλλά Επί τη ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την ψηφοφορία για το έγγραφο που νωρίτερα ψηφίσαμε για τις κατευθυντήριες γραμμές για το 2019 και με την ευκαιρία θέλω να αξιοποιήσω τη μέθοδο εργασίας την ίδια που είχαμε και για τις κατευθυντήριες γραμμές με τις ε, προπαρασκευαστικές δράσεις για τα πιλωτικά σχέδια που θα προχωρήσουν με συντονισμένη συνεργασία μεταξύ συναδέλφων και πολιτικών ομάδων ώστε να δώσουμε απαντήσεις στις ε, πολιτικές ενδείξεις της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου που προσφέρει αυτό το έγγραφο. Ο συνάρφος Μουρεσάν πέρσι ε, πραγματοποίησε εξαιρετική δουλειά για το θέμα αυτό και θα εμπνευστώ κι εγώ από, την, ε, το παράδειγμά του. Επίσης, σημειώνω ευθύς εξ αρχής ότι θα λάβουμε υπόψη και την αξιολόγηση που θα συμπεριλάβει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τις προτάσεις της για τα πιλωτικά σχέδια. Αλλά το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή μας, ολόκληρη η Ολομέλεια, έχει απόλυτη ελευθερία να αξιολογήσει τις προτάσεις δεν θα δεσμευτούμε δηλαδή από τις τεχνικού χαρακτήρα αξιολογήσεις που θα μας υποβάλει η Επιτροπή. Έτσι, η πρόθεση είναι, και θα περιμένουμε βέβαια τις ε, προτάσεις ε, των ε, συναδέλφων και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εμείς θα αξιολογήσουμε πλήρως με βάση τα τεχνικά στοιχεία που θα μας υποβληθούν και ενδελεχώς τα πιλωτικά σχέδια ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ τον ε, Γενικό Εισηγητή και δίνω το λόγο. Η Μόνικα έφυγε ο Σκιώδης. Κύριος Κόλμελ, θέλετε να μας πείτε δύο λόγια εσείς. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ σύντομα. Ευχαριστώ τον ε, εισηγητή. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο τομέας, ιδιαίτερα για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ακολουθεί μόνο την πεπατημένη, αλλά ότι κοιτάμε νέες λύσεις διαφορετικές. Όσο και αν είμαστε ικανοποιημένοι από πράγματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα, πρέπει να ε, κοιτάξουμε και εναλλακτικέ και είμαστε ικανοποιημένοι από τα όσα έχουμε δει μέχρι στιγμή. Ο κύριος Δεπρέ μας εγκατέλειψε. Α, όχι, όχι, εδώ είναι. Κύριε Δεπρέ, θέλατε εσείς να μας ε, δώστε την αξιολόγησή σας για τα πιλωτικά σχέδια προπαρασκευαστικές δράσεις. Είστε σκιώδης. Πρόεδρε δεν το είχα υπόψη μου ότι είμαι σκιώδης. Αλλά μια και ήμουν και αφηρημένος εκτός από σκιώδης. Καλώς λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ για την γνώμη σας. Κυρία Μυριάντα, δεν είστε εδώ. Τάραντ. Ας τον αφήσω. Ας τον αφήσω να τελειώσει τη του όχι, συνδιαλεξή του. Δεν θέλει. Όπως και ο κύριος Δεπρέκης. εσείς, ωραία. Ο Ζόλτεκ δεν είναι εδώ. Ωραία. Πολύ καλά πάει η έκθεσή σας κύριε. Ναι, πρόεδρε, άρα, άρα πράσινο φως για μένα και ξεκινάω τη δουλειά μου. Μα είναι πολύ σημαντικό όμως, λέει ο πρόεδρος, το θέμα σας. Γιατί είναι από τα λίγα θέματα στα οποία έχει το κοινοβούλιο περιθώριο με τις προπαρασκευαστικές δράσεις, με τα έργα αυτά, μπορούμε να επηρεάσουμε κατά κάποιο τρόπο τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι μεγάλη ικανοποίηση όταν μπορεί κανεί να προτείνει ένα δοκιμαστικό σχέδιο να το φέρει σε πέρα και βέβαια πρέπει μετά να γίνει και η αξιολόγηση του έργου αλλά και τη αποτελεσματικότητά του και αυτή θα πρέπει να γίνεται σωστά γιατί καμιά φορά έχουμε την εντύπωση πω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, κατακυριεύεται από μια αίσθηση αδράνειας δεν ξέρω τι κυρία Σαβάλ. Σάμπαλ. Ε, για τον έλεγχο, είπατε και την αποτελεσματικότητα, ναι, και την εφαρμογή την ίδια, όχι μόνο την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής. Ο κύριος Ρούμπιχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα πιλωτικά ή δοκιμαστικά έργα βεβαίως έχουν εν γέννη καινοτόμο προσέγγιση. Και είναι καλό αναλόγως να τα προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή πολύ συχνά μπορεί να αλλάζει τις προτεραιότητες. Για μας, ωστόσο, πρόκειται για ένα είδος ε, δικαιώματος πρωτοβουλίας. Μπορούμε δηλαδή έτσι, μέσω της Επιτροπής των Προϋπολογισμών, να δώσουμε όθηση στους πολίτες, εκφράζοντας κάποιες προτιμήσεις, ε, κάποιες επιθυμίες ως προς τη, τα προσυλλοποίηση έργα. Αλλά βέβαια η τελική επιλογή ανήκει στην Επιτροπή. εμείς μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι άμα δώσουμε κακή βαθμολογία βγαίνει από τον κατάλογό μας. Υπάρχει μια ισορροπία. Αλλά πρέπει και η Επιτροπή περισσότερο να ε, ακολουθεί, να υπακούει αυτά τα οποία εμείς εκ μέρους των πολιτών μας έχουμε εκφράσει ως προτιμήσεις. Κύριος Δεπρέ, Πρόεδρε, ευχαριστώ και πολύ σύντομα. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί είπατε <laughs> αυτό ακριβώς που θα μπορούσα να είχα πει εγώ. Μα εγώ σας ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Επιβεβαιώνετε τα λόγια μου. Και αν δεν κανεί το λόγο, ναι και έχουμε και τόσο χρόνο, έχουμε ήδη προχωρήσει περισσότερο, πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε την, ε, με τη διεξαγωγή της προφορίας. Θα ήθελα να πω δύο προσωπικά λόγια. Είχαμε την, ε, το δοκιμαστικό έργο για το εξάμεινο των μαθητευομένων στην κινητικότητα. Ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να πάρει το χρόνο του, να προχωρήσει και η προσαρμογή για την κινητικότητα αυτή και των εθνικών εργατικών νομοθεσιών κτλ. Όμω ήταν κάτι το οποίο εμεί είχαμε προωθήσει, η Ευρωπαϊκή Επίτροπη το δέχθηκε. Το πρικοδότησε και με 400 εκατομμύρια για την περίοδο 18 ε, με 20 χαρακτηρίζει Εράσμους Προ, επαγγελματικό Εράσμους δηλαδή, τα σχετικά προγράμματα και βάζει στην, ε, στο τραπέζι των συζητήσεων του Συμβουλίου τον Οκτώβριο ένα καταστατικό ενιαίο μια συμφωνία για καταστατικό ενιαίο των μαθητευομένων και τη, με, την προοπτική αυτή της κινητικότητας, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα η μαθητεία να εξασφαλίζεται και με ε, κινητικότητα διασυνοριακή με στόχο και την επίλυση του προβλήματος της ανεργίας των νέων κύριε Ρούμπιχ και για την Αυστρία και για τη Γερμανία και για τις κάτω χώρες έχει μεγάλη σημασία αυτό και άρα βλέπετε ότι μπορούμε χάρη σε αυτές τις πρωτοβουλίες μας να φέρνουμε ιδιαίτερη πρόοδο ίσως το προσεχές που δουπού να έχουμε ένα ιδιαίτερο ε, κεφάλαιο πρόγραμμα για την ε, μαθητεία και την κινητικότητα. Κύριε Βιώτη, Η γνώση σας και η επιμέλειά σας είναι για μας εγγύηση ότι θα προαχθούν για το 2019 τα πιο πολλά υποσχόμενα δοκιμαστικά έργα ή σχέδια. Και βεβαίως επισημαίνω τις προθεσμίες που έχουμε να σεβαστούμε. Τα σχετικά προγράμματα πρέπει στις ε, σχετικές τροπολογίες, συγγνώμη, πρέπει 27 Απριλίου να έχουν κατατεθεί, άρα έχουμε 1,5 μήνα, προτάσεις αποκλειστικά και μόνο με βάση το e-committee, το έγγραφο που έχουμε στο e-committee της Επιτροπής μας και το σχετικό σύνδεσμο τον έχετε στα έγγραφά σας επίσης. Euh, θέλει η Επιτροπή να μας δώσει κάποιες διευκρινήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιες ενδείξεις όσον αφορά αυτά τα δοκιμαστικά προγράμματα, την αξιολόγηση κλπ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευπρόσδεκτη αυτή η συζήτηση που έγινε σήμερα εδώ, η ανταλλαγή απόψεων. Κατέστη σαφές στη μεσοπρόθεσμη έκθεση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και κάποιες μέρες παρουσίασε μια πολύ καλή εικόνα όσον αφορά την υλοποίηση των 88 δοκιμαστικών αυτών προγραμμάτων και προπασκευαστικών δράσεων που περιλαμβάνονται στον προπολογισμό του 2018 και μόνο ένα από τα 88 δεν θα εφάρμοστεί. Τρία ακόμα εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ καλό αυτό λοιπόν. Είναι μια επιτυχία που αποδεικνύει την ποιότητα του επιτελεστέντος προπαρασκευαστικού έργου. Είναι δουλειά που έκανε συγητή και οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κλείνοντα, θέλω να ευχηθώ στο Γενικό Συγητή για τον προπολογισμό του 2019 ό,τι καλύτερο και διαβεβαιώνω ότι πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα του παράσχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη όπω κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν. Είχαμε άριστο ρυθμό εργασιών. Έπρεπε να ολοκληρώσουμε τις ψηφοφορίες στις 10. και να εξετάσουν σχέδιο προϋπολογισμού για το Κοινοβούλιο, έκθεση Ρούβιχ στις 10 και 4. Είμαστε μισή ώρα πιο γρήγοροι, είναι πιο νωρίς. Ο Πολ Τούμπικ. Θα έχουμε μια συνεδρία σε ανοιχτή και μια κυκλισμένη των θυρών σε δύο τμήματα. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Προπολογισμό του 2019 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, καταλαβαίνετε ότι είναι ιδιαίτερη η χρονιά αυτή. Μερικά από τα θέματα είναι καινούρια, αυτά που θα πρέπει να προσέξουμε. Είτε πρόκειται από τη μια για το Brexit, που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα το 2019, αλλά υπάρχει και το πρόγραμμα για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Για την επόμενη ετία δηλαδή η κατάρτιση του προϋπολογισμού και θα έχει επιπτώσεις. Επίση ξέρουμε ότι έχουμε και ευρωεκλογέ το 2019. Οπότε και από αυτή τη σκοπιά θα πρέπει να γίνουν απαραίτητες τροποποίησεις στον προπολογισμό του Κοινοβουλίου. Η προετοιμασία των εκλογών είναι κάτι το οποίο συναντάμε σε κάθε νομοθετική περίοδο. Έχουμε στοιχεία αριθμητικά από την προηγούμενη περίοδο τα οποία μας δείχνουν ότι οι εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν επιπτώσεις για τον προϋπολογισμό. Ε, προετοιμασία της επικοινωνίας ε, για να ενημερωθούν οι πολίτες και να ε, παροτρινθούν να ψηφίσουν έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό για το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να ενημερώνεται ο πληθυσμός όχι μόνο για τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για τα μελλοντικά του σχέδια, αλλά και για τα δικαιώματα των πολιτών που απορρέουν από τις εκλογές αυτές. Και βεβαίω τα διάφορα πολιτικά κόμματα, ποια είναι, ποιε είναι οι διάφορε ιδέε και σκέψει για το μέλλον τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Όλα αυτά θα πρέπει να τα παρουσιάζει και το Κοινοβούλιο σε ένα ευρύ ε, φάσμα και μια ευρεία πολιτική συζήτηση είναι απαραίτητη για να δείξουμε στους πολίτες, άνδρες και γυναίκες ότι εδώ Επιθυμούμε τη συνεργασία ε, στην Ευρώπη να τη βελτιώνουμε. Ποια είναι τα κέντρα βάρους της έκθεσης μου, έρχομαι τώρα στο γενικό τμήμα. Η πρόταση του Προεδρείου ε, είναι αυτή τη στιγμή στο 18,79%. Έχουμε διαβάσει στο Προεδρείο ότι το 20% είναι η κόκκινη γραμμή μας. Δηλαδή σε καμία περίπτωση το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να ξεπεράσει το 20% από το τίτλο 5 για διοικητικές δαπάνες. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που το Προεδρείο τηρεί αυτή την κόκκινη γραμμή και δεν την παραβιάζει. Αυτή που ήταν κόκκινη γραμμή και τα προηγούμενα έτη, δεν είναι τίποτα καινούριο και πόσο μάλλον του χρόνου που είναι εκλογική χρονιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συγκρατηθούν όσο γίνεται οι δαπάνες και να περικοπούν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να είναι και παράδειγμα προς μίμηση από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Γι' αυτό και η τρέχουσα πρόταση του Προεδρείου είναι στα 18,79%. Εδώ και 15 χρόνια είναι το χαμηλότερο ποσοστό αυτό που έχει προταθεί και δείχνει και την τακτική και τη λογική που μας διέπει ας προς τις περικοπές αυτές που θέλουμε να τις κάνουμε αλλά να τις συνδέσουμε και με αποτελεσματικότητα. Ε, ε, δηλαδή κυριαρχεί πάντα εδώ το στοιχείο των οικονομιών και της αποτελεσματικότητας. Ο προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυξάνεται κατά 3,9% συνολικά ε, λιγότερο από τον τίτλο 5 που αυξάνεται κατά 4,25%. Δηλαδή και εδώ βρισκόμαστε κάτω του τίτλου 5 και μπορούμε να είμαστε λίγο πιο φιδωλοί. Ε, 3,9% μπορεί να φαίνεται εκ πρώτης όψεως μεγάλη αύξηση, αλλά θα πρέπει να ειδωθεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Ότι ε, έχουμε ε, υψηλές έκτακτες δαπάνες για ε, την εκλογική χρονιά 37,3 εκατομμύρια συν 34,3 εκατομμύρια δαπάνες για την ασφάλεια και διάφορα άλλα ε, που άπτονται των εκλογών. Σύνολο 71,6 εκατομμύρια. Και ξέρουμε ότι τα δύο τρίτα του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, συνδέεται με την τη μαριθμική αναπροσαρμογή, ε, κυρίως για τους μισθούς και τις απολαβές και αποζημιώσεις βουλευτών και υπαλλήλων, αλλά και τις συμβάσεις για τα κτίρια. Ε, σε ένα γενικό πλαίσιο, λοιπόν, θα πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά και στη συζήτηση θα πιέσω να γίνουν και άλλες περικοπές και άλλες οικονομίες ε, στο προϋπολογισμό αυτό και αντίστοιχα θα χρειαστούν διαπραγματεύσεις με το Προεδρείο του Κοινοβουλίου και θα επιδείξουμε την απαραίτητη ακαμψία. Για το Brexit έχουμε ένα καλό νέο. Στις 8 Δεκεμβρίου αποφασίστηκε ο προπολογισμός του 2019 και του 2020 να θεωρεί ακόμα την ε, Μεγάλη Βρετανία κράτος μέλος. Αυτό μας δίνει ένα περιθώριο ε, σταθερότητας για το επόμενο διάστημα σχετικό. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το δημοσιονομικό πλαίσιο αφορούν όλες τις παραμέτρους του προϋπολογισμού. Για μένα είναι πολύ καλή είδηση αυτή ότι λαμβάνονται αποφάσεις προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ξέρουμε ότι υπάρχει και το ε, ε, περίφημο ζήτημα της έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Είμαστε πολλοί βουλευτές, πλειοψηφία που θέλει μια έδρα. Ε, ο καυγάς αρχίζει όταν πρέπει να αποφασιστεί ποια θα είναι αυτή η έδρα. Νομικά και νομοθετικά η έδρα μας είναι το Στρασβούργο και για να αλλάξει θα πρέπει αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων να αποφασίσουν ομόφωνα. Και όταν έχει 28 κράτη-μέλη, 27 στο μέλλον, αυτό είναι πρόκληση. Το κοινοβούλιο μπορεί να επιθυμεί ό,τι θέλει, αλλά τις αποφάσεις τις παίρνουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με το συμπληρωματικό προπολογισμό ε, στο θέμα αυτό γιατί την 1η Απριλίου με το Brexit φεύγουν οριστικά οι βουλευτές από τη Μεγάλη Βρετανία αλλά ε, και τα θεσμικά όργανα και χάνουν την ε, επίρροή τους στα υπόλοιπα κράτη-μέλη και έχει ενδιαφέρον να δούμε τον Απρίλιο του 19 ποια θα είναι η νέα σύνθεση του Κοινοβουλίου όταν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι όργανα λήψης αποφάσεων με δικαίωμα ψήφου. Προς μεγάλη μας λήψη. Έρχομαι τώρα στις εκλογές, ευρωεκλογές του 2019, που καταρχήν θα γίνουν απουσία της Μεγάλης Βρετανίας. Η Μεγάλη Βρετανία ε, απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και δεν είναι πλέον μέλος στη δημοκρατική συνεργασία. Για μας παρόλα αυτά έχει σημασία να δείξουμε ότι μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους η συνεργασία στην πολιτική μας έχει αποδείξει ότι οι πολίτες μας έκτοτε μπορούν να ζουν σε συνθήκε ειρήνη, χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ότι τα ζητήματα δεν λύνονται με στρατού, αλλά με πολιτικού που δίνουν τα χέρια και συμφιλιώνονται και ακόμα και αν έχουν χάσει μια ψηφοφορία μπορούν να πιούν ένα καφέ και να συζητήσουν το επόμενο θέμα. Δεν συμφωνώ ούτε εγώ με όλες τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φαντάζομαι κανένας από εμά δεν είναι πανευτυχής και είτε συγνωρίζουμε, αλλά αυτά έχει πολιτική ζωή. Και αυτό δείχνει όμως ότι μπορούμε να συνεργαζόμαστε χωρίς βία και με ειρήνη για να λύνουμε μεγάλα προβλήματα των πολιτών με τέτοιο τρόπο. Άρα, 33 εκατομμύρια για την προεκλογική εκστρατεία. Δεν είναι πολλά τα λεφτά. Ας σκεφτείτε ότι πρόκειται για 500 εκατομμύρια πολίτες, άνδρες και γυναίκες. Ξέρετε, γίνεται μια συζήτηση, τι αναλογεί τώρα αυτό, τι, τι αντιπροσωπεύει. Ένα καφέ, μισό καφέ, ένα πολίτη, κάτι τέτοιο, μισό καφέ α πούμε. Είναι πολύ φιδωλός ο προπολογισμό. Ξέρουμε ότι τα κόμματα στις χώρες μας, τα πολιτικά, αγωνίζονται με να κάνουν προεκλογική εκστρατεία χωρίς πόρους ή χωρίς επαρκείς οικονομικούς πόρους και ούτε ε, προσωπικό θέλουν να μας διαθέτουν για τις ευρωεκλογέ. Και ό,τι αφορά λοιπόν τα ευρωπαϊκά θέματα, ε, προσκλούει στην απροθυμία των κομμάτων να βοηθήσουν. Οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει και γραφεία ενημέρωση και τη διαδικασία του κορυφαίου επικεφαλής του ψηφοδελτίου του Candidates. Οπότε μπορούμε να δημορφώνουμε την πολιτική μας με ανοιχτές εκλογές, με δημοκρατικές εκλογές. 50% περίπου των βουλευτών δεν κατέρχονται ξανά υποψήφοι ή δεν επανεκλέγονται. Οπότε ε, ε, υπάρχει συνέπεια και για τον προπολογισμό. Οι απερχόμενοι βουλευτές, οι βοηθοί τους, οι σταζιέρ τους, ε, θα πρέπει να λάβουν κάποια αποζημίωση. Εγγράφεται αυτός ο προπολογισμό, ο ΕΦΑΠΑΞ, για τη συγκεκριμένη εκλογική χρονιά και βεβαίως και οι Βρετανοί βουλευτές θα πάρουν αυτή τη μεταβατική προσωρινή αποζημίωση υποχρέωση είναι ε, εγγυημένη μέχρι το 2020. Το επόμενο μέγα ζήτημα είναι η μεγάλη ιστορία της ασφάλειας και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αποφασιστικό, γιατί είχαμε κάποιο επεισόδιο όχι μόνο στο Βέλγιο, αλλά και περισσότερο διαπιστώνεται βίαιη συμπεριφορά και θα πρέπει αντίστοιχα να θωρακίζουμε αφενός τα κτίρια μας, αφετέρου να τα αφήνουμε όσο γίνεται ε, προσβάσιμα στους πολίτες. Στις εισόδους έχουν περίπου ολοκληρωθεί εργασίες και είσοδος για τους επισκέπτες. Έχουμε τον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, έχουμε το Παρλαμεντάριο. Είναι ελκυστική η προσφορά για τους επισκέπτες και στο Στρασβούργο διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο για τους επισκέπτες, ε, μια διαδρομή για να καταλαβαίνουν καλύτερα πώς λειτουργεί η δημοκρατία στην Ευρώπη. Υπάρχουν κάποια πρακτικά παραδείγματα ε, πάρα πολύ ε, εύχριστα και παραστατικά που επιτρέπουν στους επισκέπτες να δουν πώς δουλεύουν οι βουλευτές. και όπως σε κάθε σχολείο ή σε κάθε επιχείρηση δεν είναι πάντα παρόντες στην Ολομέλεια βουλευτές για να δείχνουν παρουσία. Έχουν και άλλες δουλειές ταυτόχρονα. Και από τους επιτρόπους δεν είναι και 28 παρόντες, είναι ένας κατά κανόνα που είναι αρμόδιος για το θέμα και οι λίγοι βουλευτές που είναι επίσης αρμόδιοι και έχουν να μιλήσουν. Οι συζητήσεις εντατικές γίνονται στις πολιτικές ομάδες και στις επιτροπές. Και αυτά τους εξηγούμε για να καταλαβαίνουν οι επισκέπτες τι βλέπουν και τι γίνεται. Είναι πολύ σημαντικά για μας. Θα συνεχίσουμε και το πρόγραμμα δράσης για την κυβερνοασφάλεια, εξασφάλιση των επικοινωνιών και αποτελεσματικότητα θα πρέπει να έρθει στο προσκήνιο. Και επίσης η επικοινωνία ε, και η ενημέρωση του κοινού είναι πάρα πολύ σημαντική Έχουμε 800 τριμερείς διαλόγους ε, σε αυτή τη θητεία και έκτακτες επιτροπές, οι οποίες πολλαπλασιάζονται συνεχώς. Και θα παρακαλούσα τους συναδέλφους να φροντίσουν αυτές οι έκτακτες επιτροπές μάλλον να καταλάβουν οι συνάδελφοι ότι αυτές οι έκτακτες επιτροπές επιβαρύνουν σημαντικά τον προπολογισμό. Έχουμε μετατάξεις εκεί, αποσπάσεις υπαλλήλων, επιπλέον κόστος για τη διερμηνία. Με αυτές τις έκτακτες επιτροπές που συστήνονται, χάνουν προσωπικό οι τακτικές μόνιμες επιτροπές και όχι μόνο υπαλλήλους αλλά και δυνατότητα συνεδριάσεων ε, χρονική θα πρέπει η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών να αποφασίζει ποια είναι η Ενική Επιτροπή, η Διαρκή Τακτική Επιτροπή του Κοινοβουλίου που είναι αρμόδια για το συγκεκριμένο θέμα και να γίνεται εκεί η δουλειά και όχι σε έκτακτη επιτροπή κάθε φορά. Έχουμε επιτροπές Εκεί θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλές οικονομίες και ε, όχι μόνο χρημάτων αλλά και κόπου και διοικητικέ. Γιατί δεν είναι νομοθετική η δουλειά που κάνουν αυτές οι επιτροπές. Θα είχε νόημα λοιπόν. Έρχομαι στο επόμενο θέμα που είναι τα κτίρια. Η Μόνικα Χόλμαϊερ μας τα είπε αυτά ήδη. Για το κτίριο Αντεναόερ για παράδειγμα στο Λουξεμβούργο η Ανατολική Πτέρυγα θα είναι έτοιμη ε, το 2018 για παραλαβή. Θα δούμε η Δυτική το 2019 και βλέπουμε. Η χρηματοδότηση του κτηρίου Κόρατ Αντενάουερ ΚΑΤ νομίζω έγινε με τρόπο πάρα πολύ διαφανή και θα πρέπει μάλλον να γίνει αυτό Θέλουμε περισσότερες λεπτομέρειες και τις ε, λάβαμε από το Προεδρείο ε, για το πόσο απέχει η επιθυμητή ε, κατάσταση από την πραγματικότητα και ποια πράγματα παραμένουν ακόμα εκρεμή μέχρι να είναι έτοιμο το κτίριο για παράδοση, για παραλαβή από εμά και να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τι δημοσιονομικές συνέπειες θα έχει για μας. Ξέρουμε και τη συζήτηση που γίνεται ε, για την Ολομέλεια, ε, για το, το κύκλιο στις και στο Στρασβούργο, την αίθουσα της ολομέλεια. Και στις δύο αίθουσε έχουν ανακαινιστεί ε, οι οροφές. Θυμάμαι κάτι συγκλονιστικές φωτογραφίες όπου είχε πέσει ένα δοκάρι και κατέστρεψε τη δική μου, το δικό μου έδρανο και κάποιων γειτόνων. Ευτυχώ που έγινε καλοκαίρι, θα είχαμε δράματα. Ε, οπότε η ασφάλεια των κτίριων τίθεται. Δεν είναι μόνο θερμικές εκεί οι εντάσεις, <laughs> υπάρχουν και άλλες εντάσεις που πλήττουν τα κτίρια και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα και για την ασφάλεια των επισκεπτών, των εργαζομένων, των βουλευτών. Ε, αυτό είναι θέματα προτεραιότητας. Άρα δεν θα πρέπει να κάνουμε έτσι μια βραχυπρόθεσμη ανακαίνιση, αλλά και μεσοπρόθεσμα να δούμε ποιε είναι οι κτηριακές μας ανάγκες και υποχρεώσεις ε, και ε, οι εργασίες, οι κοινοβουλευτικές έχουν αλλάξει πολύ το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια και θα πρέπει αυτό να ανακλάται και στα κτίρια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τους συνεργάτες ε, των βουλευτών, τους βοηθούς τους να έχουν αξιοπρεπή γραφεία με συνθήκες εργασίας όπως φαντάζεται κανείς και από κοινωνική σκοπιά. Αυτή τη στιγμή έχουμε στις Βρυξέλλες ένα συν δύο γραφεία και στο Στρασβούργο ένα συν ένα. Και ο εξοπλισμός των γραφείων για την επόμενη περίοδο θα είναι σημαντική γιατί έχουμε μια νέα γενιά βουλευτών που θα μας έρθει οι οποίοι στον τομέα της πληροφορίας και της επικοινωνίας έχουν και νέες απαιτήσει ε, που θα προβάλλουν στο Κοινοβούλιο. Βλέπουμε εδώ που καθόμαστε ούτε μπρίζες δεν έχουμε στα έδρανά μας ναι. για να φορτίζουμε τις συσκευές. Πόσο μάλλον, πόσο μάλλον το διαδίκτυο και η ποιότητα του ίντερνετ ε, στο Κοινοβούλιο. Χωράει πολύ η βελτίωση. Ε, λοιπόν, τώρα συντομεύω. Βεβαίως θέλουμε να συνεχιστεί το one-stop shop για τους ε, διαπιστευμένους ε, βοηθούς, να συνεχίσει το καθεστώς των βουλευτών, λιγότερη γραφειοκρατία και για τους βουλευτές και για τους βοηθούς, μείωση των γραπτών υποχρεώσεων. Έχουμε πολλές συμβάσεις τώρα και πολλές διατυπώσεις και αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο για τη διεκπαιρέωση διαφόρων διοικητικών και γραφειοκρατικών ε, ζητημάτων. Να το ξανασκεφτούμε αυτό παρακαλώ για να δούμε πώς μπορούμε να το απλουστεύσουμε. Προσωπικό. Έχουμε κάνει οικονομίες 59 ε, θέσεις, ε, έχουμε μειώσει κατά 1% ε, το χρόνο ε, το προσωπικό και φτάσαμε στο στόχο του 5% στην πενταετία. Ελπίζω και τα κράτη-μέλη να το λάβουν αυτό υπόψη και να το ακολουθήσουν για να έχουμε καλύτερη λειτουργία. Τελειώνω. Χρονοδιάγραμμα. Μέχρι τις 14 Μαρτίου μπορείτε να καταθέσετε τροπολογίες και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 ε, του μηνός θα συζητήσουμε τις τροπολογίες εδώ με χαρά και ήδη χαίρομαι για τα σχόλια των συναδέλφων που θα ακούσουμε στη συνέχεια για να μπορέσουμε να ε, έχουμε μια αποτελεσματική έκθεση και χρήσιμη για την κοινή γνώμη όσο γίνεται καλύτερα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Merci, Σας ευχαριστώ κύριε Σιγητά για την παρουσίαση του σχεδίου εκθέσεώς σας. Όσον αφορά τον ενδεχόν προπολογισμό του Κοινοβουλίου του 2019, κάτι έκτακτο εξαιρετικό, διότι αφορά και την ανανέωση της θητείας του Κοινοβουλίου. Την ανανέωση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ για όλες τις διευκρινήσεις που κάνατε. Θα καλέσω τους και τους συγητές να εκφράσουν την άποψή τους. Η κυρία Γκαδίου Ζαμπάλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω διάφορα σχόλια να κάνω και μία παράκληση. Να αρχίσω από την παράκληση. Ο κύριος Ρουμπίχ και οι υπόλοιποι σκιώδες ε, εργαζόμαστε χωρίς να έχουμε επίσημη ενημέρωση για το τι θα εγκρίνει το Προεδρείο. Γιατί ξέρετε ποιες είναι οι προθεσμίες στο Προεδρείο και τελικά το μόνο επίσημο που γνωρίζουμε είναι μια προφορική ενημέρωση την περασμένη εβδομάδα. Ε, αυτά δεν είναι σοβαρή μέθοδος εργασίας και πολλά τα μαθαίνουμε ε, έτσι από το πολιστικό αισθητήριο που έχουμε και την όσφρησή μας ε, και από εμπειρία προηγουμένων ετών. Θέλω να, εκφράσω αυτή την, το παράπονο μάλλον, δεν ήταν παράκληση παράπονο, καταγγελία πιο πολύ. Όπως όλοι οι προϋπολογισμοί τέλους θητείας έχουμε έκτακτες δαπάνες λόγω της προεκλογικής εκστρατείας και λόγω της αλλαγής κοινοβουλευτικής περίοδου. Φεύγουν βουλευτές, συνεργάτες, έρχονται άλλοι, χρειάζονται ε, να προβλέψουμε έκτακτες δαπάνες. Αυτό είναι αναπόφευκτο, είναι μοιραίο. Και επίσης τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει πάρα πολλές επενδύσεις στην ασφάλεια. Ε, που ενέκρινε το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας. Άρα θα συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε αυτά τα οποία έχουμε εγκρίνει για την ασφάλεια. Όπως είπε ο κύριος Ρουβίχ και το λέει και στην έκθεσή του και στην πρότασή του, προσπαθούμε πάντα να συγκρατούμε τα έξοδα. Και η καθημερινή δουλειά και οι δαπάνες να μην αυξάνονται πάνω από τον τιμάριθμο. Και πολιτικές ομάδες θα πρέπει να δουν που μπορούν να κάνουν περικοπές για να ε, μην ξεπερνάνε τον τιμάριθμο. Έχουμε ένα άλλο πρόβλημα που βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Το Προεδρείο παίρνει πολλές αποφάσεις που έχουν δημοσιονομικές συνέπειες χωρίς να έχουμε εμείς εγκρίνει τίποτα, ούτε καν έχουμε συμμετάσχει στη λήψη των αποφάσεων. Για παράδειγμα, αποφάσισε το Προεδρείο να αλλάξουν τα γραφεία στο Στρασβούργο και να αυξηθεί ο χώρος που έχουμε. Νομίζω ότι υπάρχουν και προτάσεις ε, για να ανακαινιστούν τα εστιατόρια κλπ. Ωραίε αποφάσεις παίρνουν. εμεί τι εγκρίναμε. Μπορεί να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε. Αλλά ποιο μα ρώτησε. Οι λιμένες αποφάσεις έρχονται και μας υποχρεώνουν να εγγράψουμε αυτές τις δαπάνες στον προπολογισμό του Κοινοβουλίου. Και αυτή είναι η δυσλειτουργία που εμείς είχαμε εντοπίσει και προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια να διευκρινίσουμε και να ξεκαθαρίσουμε. Γιατί έχουμε και εμεί αρμοδιότητα εκεί για τη λήψη των αποφάσεων ε, και τελικά μας έρχονται αποφάσεις και θα πρέπει εμείς να τα λουστούμε. Και χωρίς να έχουμε επίσημη ε, πληροφόρηση, προεξοφλώ ότι θα κάνουμε προτάσεις σε διάφορα θέματα. Ένα θέμα που ήταν αρκετά επίμαχο στην Επιτροπή μας και προσπαθήσαμε και τα τελευταία χρόνια να αντιμετωπίσουμε ήταν τα γενικά έξοδα Ακριβώ επειδή δεν υπήρχε νέα πρόταση από το Προεδρείο, που υποτίθεται ότι δουλεύουν την πρόταση αυτή αυτά τα χρόνια, καταφέραμε να συμφωνήσουμε για μια παράγραφο που ε, αντανακλούσε την αίσθηση της πλειονότητας των βουλευτών και σε αυτή τη γραμμή κινούμαστε. Θα κάνουμε επίσης πρόταση για την επιστροφή ε, των εξόδων ε, αποστολών ε, των κοινοβουλευτικών ε, βοηθών. Για το 2018 ζητήσαμε να ευθυγραμμιστούν, να εξισωθούν με τις δαπάνες οι οποίες επιστρέφονται στους υπαλλήλους των πολιτικών ομάδων. Αυτό μεν εγκρίθηκε, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Δεν ξέρω αν είναι δικαιολογία ή πραγματικότητα αυτό που μας λένε, ότι Ε, δεν υπήρχε περιθώριο, ότι ήδη είχαν ε, μοιραστεί τα λεφτά. Τώρα μιλάμε για την επόμενη θητεία. Ωραία. Να δούμε από εδώ και πέρα τι θα κάνουμε. Είναι λογικό να εξισώσουμε αυτά που ισχύουν για τους υπαλλήλους των ομάδων με τους βοηθούς. Και μια που μιλάω και για δαπάνες, για την κοινοβουλευτική επικούρηση, σε αυτό το σχέδιο έκθεσης προτείνεται να αυξηθεί αντίστοιχα μια εύλογη αύξηση νομίζω. Σοσιαλιστική ομάδα είχε ζητήσει να υπάρξει αύξηση στην αρχή της θητείας για διάφορους λόγους και αν διατηρηθεί όμως η σημερινή κατάσταση θα πρέπει να είναι αρκετά ε, ικανοποιητική για να ε, έχουμε και αξιοπρεπείς μισθούς για τους εργαζομένους στο Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια, τι γίνεται με τις προϋποθέσεις για τους ε, υποτρόφους και τους στασγέρ μάλλον τους ασκούμενους στο κοινοβούλιο. Το έχουμε μελετήσει σε μια ομάδα εργασίας. Δεν είναι ικανοποιητική η κατάσταση. Κάναμε μια μικρή έρευνα και διαπιστώσαμε ότι γύρω στο 20% το 1 πέμπτο των ασκουμένων των σταζιέρ έχουν ένα μισθό γύρω στα 1000 ευρώ. Θα πρέπει όλοι, ανεξαιρέτως όσοι εργάζονται σε γραφείο βουλευτών, πολιτικές ομάδες και στη διοίκηση ως ασκούμενοι θα πρέπει να έχουν αξιοπρεπή μισθό. Όπως στην Κομισιόν. Και όχι μόνο μισθό, θα πρέπει να έχουν και κοινωνική ασφάλιση, ε, τη βασική, και ένα σχέδιο ε, για εκ, εκπαίδευσή τους. Γι' αυτό είναι και υπότροφοι, ας πούμε, και σταζιέρ. Εμείς βγαίνουμε και τα πετούμε όλα αυτά από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ε, να μην ε, κακοποιούν και να μην στραπατσάρουν αυτό το θεσμό του ασκούμενου. Και θα πρέπει να το είδα να κάνει και το Κοινοβούλιο και να ζητήσουμε από το Προεδρείο να έχουν κάποιους ε, όρους και ελάχιστες προϋποθέσεις στις συμβάσεις που υπογράφονται με τους ασκουμένους. Αυτά. Και χωρίς πληροφόρηση. Εν πάση περιπτώσει, εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόλμελ έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή μας ότι αυτά που μας είπε όχι μόνο ήταν, μας έδωσαν μια πλήρη επισκόπηση, αλλά ήταν και τόσο λεπτομερή στοιχεία όσο πράγματι χρειαζόμαστε. Και θα συμφωνήσω με τη συνάδελφο Καρδιά Σοβάλ ότι πρέπει να κοιτάξουμε να έχουμε τα ακριβή αριθμητικά στοιχεία ώστε να μπορούμε να μιλούμε με στοιχεία. Εν όλο όμως η βασική γραμμή που μας προτείνει ο εισηγητής είναι απόλυτα ικανοποιητική για μας. Είναι σωστό καταρχάς ο σχεδιασμός να γίνει με τους 751 βουλευτές, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει, εφόσον πρόκειται βέβαια να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών με την ολοκλήρωση του Brexit, θα δούμε τι θα κάνουμε. Πάντως ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει με μεγάλη διαφάνεια, ώστε να μην δοθεί εντύπωση ότι δημιουργήθηκε ένα αποθεματικό το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί κανείς να ε, χρησιμοποιήσει μεταθέτοντάς το σε άλλες δαπάνες. Θα πρέπει αυτό να γίνει με απόλυτη διαφάνεια λοιπόν και σε ένα έτος εκλογικό έχει τεράστια σημασία η διαφάνεια. Επίσης τεράστια σημασία έχει, όπως ακούσαμε ήδη άλλωστε, να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις ειδικότερα να έχουμε ικανούς υπαλλήλους προσωπικό με δεξιότητες όλο και περισσότερο απαιτητικά είναι, όλο και περισσότερο απαιτητική είναι η εποχή στην οποία ζούμε. Χρειάζεται κανείς στην ομάδα του να έχει ανθρώπους που είναι ικανοί να καταλήξουν σε μια συμφωνία να κάνουν μια δουλειά, αλλά χρειάζεται και η τεχνική, χρειάζονται και οι τεχνικές υποδομές. Δεν πρέπει να λησμονούμε και αυτό, πρέπει να δώσουμε κάποια... να δώσουμε και την ε, υποστήριξη τεχνική με την πληροφορική. Και έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Βεβαίως έχω εμπιστοσύνη στη διοίκησή μας Ιδιαίτερα όμως πρέπει, και το έχουμε πει πολλές φορές, να μειωθεί η γραφειοκρατία. Μπορεί να ακούγεται πολύ συχνά αυτή η φράση, αλλά πρέπει πια σοβαρά να την αντιμετωπίσουμε. Η επέκταση της ε, γραφειοκρατίας οπωσδήποτε απορροφά κονδύλια του φορολογούμενου. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί όταν κάνουμε πολύ λεπτομερείς τους κανόνες ασφαλώς γίνονται και πιο περιπλοκή διαχείρισή τους και γι' αυτό θα ήθελα να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί κάθε χρόνο είναι και πιο δύσκολη η υλοποίηση των δεσμεύσεων και βέβαια εάν κάνουμε ε, τόσο λεπτομερείς τους κανόνες ώστε να απαιτείται παραδείγματι να μετράμε με το χάρακα ε, το μέγεθος των λογοτύπων των ε, ομάδων, τότε βεβαίως θα χρειαστούν και παραπάνω υπάλληλοι θα επεκταθεί η γραφειοκρατία. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε θέση να μετράμε την ε, ε, επέκταση της γραφειοκρατίας με αυτόν τον όρο. Ε, πρέπει ανάλογα με το μέγεθος, με τον όγκο μάλλον της χρηματοδότησης να ορίζεται και η διαδικασία με βάση την οποία γίνεται μία σύμβαση για προμήθεια. Ε, ναι, αλλά αυτά τα πράγματα δεν διευκολύνουν πάντα τη δουλειά μας. Πρέπει εμείς να έχουμε πάντα υποδειγματική βέβαια συμπεριφορά αλλά και να μειώσουμε τη γραφειοκρατική επιβάρυνση. Γιατί βέβαια δεν είναι δυνατόν να ορίζεται το κάθε τι στην παραμικρή του λεπτομέρεια. Ευχαριστώ. Σαν νομοθέτες, εμείς οι ίδιοι, πρέπει να κάνουμε μια αυτοκριτική, να εξετάσουμε την συνείδησή μας. Μήπως καμιά φορά μέσω τροπολογιών, μήπως και εμείς δεν συμβάλλουμε στο να περιπλέκουμε τους κανόνες. Καμιά φορά ενεργούμε την περιπλοκότητα, με κάθε καλή πρόθεση βέβαια. Το αποτέλεσμα όμως είναι δημοσιονομικοί κανονισμοί, διατάξεις, των οποίων ο περίπλοκος χαρακτήρας ε, δεν πάβει να αυξάνεται. Ευχαριστώ κύριε Κόλμελ. Ο κύριος Αλή έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Ρούμπικ. Είναι πληρέστατη η έκθεσή του Βέβαια θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε διαφορετική προσέγγιση για τη σύνταξη της εκθέσεως. Θα μπορούσε να είναι και ε, ρεαλιστική και πιο λιγότερο ρεαλιστική. Αυτή είναι ρεαλιστική. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι εδώ έχουμε εξουσία νομοθετική και θα κάνουμε διάκριση μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν θεωρώ ότι καλύπτει το πλαίσιο του Ευρωκοινοβουλίου έκθεση και τον προπολογισμό του Ευρωκοινοβουλίου για το επόμενο έτος και παρουσιάζονται σωστά τα στοιχεία. Δίνει τις αναγκαίες πληροφορίες για διάφορα γεγονότα του 19 και εκδηλώσεις λόγω των αναμενωμένων ευρωεκλογών και της διαδικασίας του Brexit για την πρόβλεψη και το πώς επηρεάζονται από αυτά τα οικονομικά του Κοινοβουλίου. Έχουμε υπόψη ότι κυρίως οι δαπάνες του προπολογισμού ε, ε, ακολουθούν και τις οικονομικές εξελίξεις, την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και σχετίζονται και τα οι δαπάνες και με τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός προπολογισμός του 2019 ε, έχει σωστή προσέγγιση παραμένει κάτω από το 20% του γενικού διοικητικού, του προπολογισμού για τα διοικητικά της Ένωσης. Αυξάνεται κατά 3,9% ο προπολογισμό εν συγκρίση με τον προηγούμενο χρόνο. Αυτό δικαιολογείται. Σχετικά με αυτό, λαμβάνουμε υπόψη κάτι άλλο. Συγκρίνοντας το ετήσιο ποσοστό αυξήσεως του προπολογισμού του Κοινοβουλίου, τελευταία πενταετία, στα πλαίσια του κατηγορίας 5, βλέπουμε ότι η αύξηση είναι μικρότερη. Καλή η ενίσχυση του διαλόγου Ευρωκοινοβουλίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτό ωφελεί τη διαφάνεια. Την καλύτερη κατανόηση του νομοθετικού έργου που επιτελείται εδώ από τους Ευρωπαίους πολίτες έχοντας υπόψη και τις επικείμενες ευρωεκλογές. Ο προπολογισμό βασίζεται στι επιδόσει. Αυτό αναφέρει η έκθεση. Αυτό είναι σημαντικό για αύξηση αποτελεσματικότητα τη απόδοση και των αποτελεσμάτων από το έργο του προσωπικού. Κυρίω στα πλαίσια των ε, προκλήσεων που μας περιμένουν ε, τον επόμενο χρόνο. Ευχαριστώ κύριε Αλή. Ο κ. Σταόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ρούμπιχ που κάνατε την όλη προσπάθεια για τον προπολογισμό. Πολύ καλή συνεργασία μας πάνω σε αυτό. Τρία σχόλια έχω. Έχουμε την ε, εξαρτία την ενημέρωση για τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τους θεσμούς πριν τις εκλογές. Κάποιες πολιτικές δυνάμεις θα επικρίνουν αυτή την προσέγγιση. Να ξανασκεφτούμε το πώς το Brexit θα επηρεάσει το Κοινοβούλιο όχι μόνο που θα χάσουμε τους καλούς Βρετανούς συναδέλφους από διάφορες πολιτικές ομάδες, αλλά θεωρώ ότι έχουμε το δυσχερέστατο πρόβλημα της χρήσης της αγγλικής γλώσσης. Και αυτό ίσως δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά την Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης. Θα γίνουν παράνομα τα αγγλικά κατά την άποψή μου. Αποφασίσαμε ότι θα εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε αυτή τη γλώσσα. Πρέπει να το ξανασκεφτούμε όμως αυτό. Τρίτον, χαίρομαι που η ΣΥγητή ακολούθησε εκ νέου την προσέγγιση συνεργασίας μεταξύ Επιτροπής Περιφερειών Κοινοβουλίου και, και της Κοινωνικής και Οικονομικής Επιτροπής. Και θεωρεί ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε επίπεδο πολλών υπηρεσιών και ο Γενικός Γραμματέας ε, ανταποκρίθηκε σε αυτή την προσέγγιση. Τέλος. Ίσως και κλεισμένο των θυρών να το συζητήσουμε αυτό που θέλω να αναφέρω. Έχουμε το θέμα του εθελοντικού συνταξιωτικού ταμείου. Πρέπει να εξετάσουμε ίσως κάθε τεχνική και νομική πτυχή. Πώς αυτό δεν θα αποτελέσει ένα άχθος για τον προπολογισμό μας ίσως δεν είναι τόσο μεγάλο το οικονομικό βάρος. Πρέπει να δούμε πώς κινήθηκαν οι προηγούμενες γενιές και ίσως αυτό να δημιουργήσει πρόβλημα για μας, έχοντας υπόψη ότι επίκυνται και οι εκλογές του χρόνου. Ευχαριστώ εκ νέου. Αυτά ήταν όλα όσα είχα να σας πω. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε ο Μάρκο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Για το σχέδιο του. Κάποια σχόλια θα κάνω και βεβαίως θα συνεργαστούμε. στο πλαίσιο της συνεργασίας εισηγητικής και οδών. Ένα θα ήθελα να σχολιάσω ξεκινώντας ε, τις επικρίσεις της συναδέλφου Γκαρδία Ζαβάλη για την απουσία εγγράφων ήδη. Πρόκειται για ένα θέμα περιπλοκό στο Κοινοβούλιο, πολιτικά αλλά και τεχνικά. Τον εργαζόμαστε χωρίς έγγραφα. Μας δυσκολεύει ιδιαίτερα, κυρίως ε, εμάς είμαστε μια μικρή ομάδα και δεν έχουμε πρόσβαση στο Προεδρείο, καθώς δεν ε, έχουμε εκεί εκπρόσωπό μας. Έτσι λοιπόν ο Πρόεδρος και ο εισηγητής ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν ταχύτατα να ασκήσουν πιέσεις για να μας χορηγηθεί η απαραίτητη ε, τεκμηρίωση απαραίτητη για να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Εν γέννη για τον προπολογισμό και σε όρους αριθμητικούς ένα σχόλιο. Πρόκειται για έναν προπολογισμό ο οποίο έχει καταρτιστεί με κοινοβούλιο με την υπόθεση των 751 μελών. Δεν ξέρουμε όμω ακόμα ποια θα είναι η κατάσταση το 2019 μετά το Brexit και την απόφαση που θα λάβει εν προκειμένου το Συμβούλιο. Έχουμε μία πρόταση πάντως της ΑΦΚΟ αν δεν απατώμε που προτείνει 705 βουλευτές για την προσεχή ε, θητεία. Άρα ενώ κάνουμε υπόθεση ε, προϋπολογισμού με 751 βουλευτές θα έχουμε λιγότερους στην προσεχή θητεία μετά τις ευρωεκλογές. Και έχουμε μια συζήτηση με ένα 3,9% σε σχέση με το 2018. Τι θα κάνουμε εάν μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών γιατί η αύξηση ε, αναλογική προς όλες τις κατευθύνσεις, το like for like δηλαδή, όπως λέγεται στα αγγλικά, ε, αλλάζει πολλά σαν αποτέλεσμα στο, στην υπόθεση των 705 βουλευτών. Και επίσης, Νομίζω ότι είναι κάπως παρακινδυνευμένη η σύγκριση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε να κάνουμε με δύο θεσμικά όργανα με διαφορετικές αρμοδιότητες. Όσοι από εμάς είχαμε και την ευκαιρία να επισκεφθούμε το Κογκρέσο, το γνωρίζουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήταν η σύγκριση αυτή αβάσιμη και θα πρέπει να την αποφύγουμε. Για τους ασκουμένους συμφωνώ με τα όσα είπε η συνάδελφος, αλλά θέλω να επισημάνω και τα εξής. Έχουμε καθήκον εμείς ως εκπρόσωποι των πολιτών να εξασφαλίσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όσους εργάζονται για μας και ενδεχομένως έχουν να πληρώσουν ε, και, το κόστος διαβίωσης, ενίκια κτλ. εδώ στις Βρυξέλλες. Βλέπουμε λοιπόν τα ζητήματα. Δυστυχώς πρέπει να ορίζουμε ένα ελάχιστο όριο, είτε το πούμε μισθό, είτε το πούμε αποζημίωση, δεν έχει σημασία, ε, ως κονδύλιο που θα χορηγήσουμε σε αυτούς ε, τους ανθρώπους που εργάζονται για μας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει μια παρέμβαση σε επίπεδο κοινοβουλευτικό, ώστε για όσους δουλεύουν για μας να προσφέρουμε αξιοπρεπή μισθό. Επίσης, πολύ συχνά ακούμε να λέγεται ότι είναι έκτακτος ο προϋπολογισμός ο οποίος ε, καταρτίζεται για το έτος των ευρωεκλογών. Δεν συμφωνώ όμως εγώ σε αυτό. Ξέρουμε ότι έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά το Ευρωπαϊκό από τα Εθνικά Κοινοβούλιο κοινοβούλια ε, έρχονται κάθε πέντε χρόνια οι εκλογές σταθερά. Επομένως το να μιλάμε για έκτακτα έξοδα σε ένα έτος εκλογών είναι σαν να μειώνουμε και τη δυνατότητά μας εμάς της Επιτροπής των Προϋπολογισμών να σχεδιάζουμε και να προγραμματίζουμε. Πρέπει να είμαστε σε θέση να προβλέπουμε, να σχεδιάζουμε εν ε, αναμονή και προβολή του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για το έτος των ευρωεκλογών πρέπει να είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό. Να υπολογίσουμε και το κόστος της ε, προεκλογικής εκστρατείας κτλ. Άρα η έννοια των έκτακτων ε, δαπανών ε, βεβαίως δεχόμενος ότι υπάρχει το Brexit και άλλα έκτακτα περιστατικά και μπορεί κάποια χαρακτηριστικά να δημιουργούν προβλήματα αλλά η, έννοια των, έκτακτο, του, του, των έκτακτων χαρακτηριστικών του έτους αυτού ε, δεν με βρίσκει σύμφωνο. Θεωρώ ότι έχουμε πολλά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαμε να προβλέπουμε ε, παγίως. Και επίσης ε, η απόφαση Προεδρείου και Γενικού Γραμματέα για αυτού τύπου τις δαπάνες επιβεβαιώνει τη δική μου την ε, θέση ότι είναι ουδέτερα δημοσιονομικά τα έξοδα για την προεκλογική εκστρατεία. Με την έννοια ότι καθιστούν σαφές στον πολίτη το πώς λειτουργεί το κοινοβούλιο, συμβάλλουν με τον τρόπο αυτό, αλλά από την άλλη βλέπω ότι μπορεί τα έξοδα αυτά στόχο ε, μπορεί να έχουν ε, στόχο να στηρίξουν μόνο κόμματα που υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέραν του ορισμού αυτής της έννοιας, ποια είναι τα κόμματα αυτά, δεν είναι σαφές για μένα, οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να θεωρηθούν πολιτικά ουδέτερες, δεν μπορούν να ε, δίνουν... υποστήριξη σε κάποια κόμματα και όχι σε άλλα. Γιατί η καθήκον του Κοινοβουλίου με την προκλογική εκστρατεία είναι μόνο να εξηγήσει πώς λειτουργεί το θεσμικό όργανο ή ως θεσμικό όργανο, όχι όμως να κάνει πολιτικές επιλογές ή να εισέρχεται στον πολιτικό, στην, σε μια πολιτική τοποθέτηση ενώπιση των ευρωεκλογών. Ε, για την κτηριακή πολιτική πάλι νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Πριν να γίνω βουλευτής, είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ και να προσφέρω συμβουλές σε διάφορα ε, ιδρύματα που έχουν να κάνουν με κτηριακή και κατασκευαστική δραστηριότητα. Νομίζω ότι με αυτά που βλέπω, εάν ήταν να κάνω επενδύσεις σε κτίρια, εγώ θα ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτικός. Η επιλογή, παραδείγματι, του γραφείου στο Παρίσι, σε έναν από τους ε, πιο ακριβούς όσο και ωραίους δρόμους των Παρισίων. μου να πολλές αμφιβολίες. Όντως είναι σωστά δαπανημένα τα χρήματα αυτά. Ήτανε το μίστομα το σωστό για το δρόμο, για το δρόμο αυτόν, για το γραφείο που βρίσκεται σε αυτό το δρόμο. Μήπως δηλαδή έπρεπε να φροντίσουμε οι πόροι αυτοί αντί να δίνονται σε ε, εντυπωσιακά κτίρια, σε ε, μεγάλους δρόμους, ε, να πηγαίνανε σε έναν αξιοπρεπή μισθό για τους συνεργάτες μας και τους ασκουμένους. Και μετά νομίζω ότι μπορούμε να βαθύνουμε στα θέματα τα υπόλοιπα κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζάνη. Ακούσαμε τους κοιόδης ηγητές μας. Τώρα στους συναδέλφους θα δώσουμε το λόγο. Ο κύριος Μακά έχει το λόγο. Που κάνει το σχετισμό μεταξύ Προεδρείου και Επιτροπής Προλογισμών. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον κύριο Ρούμπικ έξοχη δουλειά που έκανε και συμφωνώ αυτά που υπόθηκαν τον κύριο Χάιντερ που Αναφέρθηκε στην πρόσβαση στα έγγραφα και που είναι δύσκολη και είναι δύσκολο να εργαστούμε χωρίς έγγραφα, κυρίως για την ενημέρωση. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί το σύστημα. Πρόεδρε, να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Ξεκινώ από ένα πρόβλημα που προσπαθούμε να επιλύσουμε. Τα προηγούμενα χρόνια η Επιτροπή Ομόφων έχει εγκρίνει και με μεγάλη πλειοψηφία στην Ολομέλεια είχε εγκριθεί το ότι μια φορά κάθε πέντε χρόνια θα κάνει ε, προσαρμογή ε, στα οικονομικά του Κοινοβούλιο, θα κάνει τον προπολογισμό λαμβάνοντα υπόψη και τα συγκεκριμένα ε, συγκεκριμένες ανάγκες που έχουμε. θέτουμε ερωτήσεις, θέσαμε ερωτήσει στην Επιτροπή που ένα χρόνο έδωσε 10 εκατομμύρια, την άλλη 5 εκατομμύρια. Έγινε μια μειώση, μετά έγινε ε, τη μαριθμική προσαρμογή έχουμε 70 με 80 ε, ευρώ παραπάνω ε, μέσω της ανασαπροσαρμογής. Πρέπει να κάνουμε ανάλυση για να δούμε τα χρήματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τα κτίρια της αύξησης εάν επεξεργαστούν σαν τον προπολογισμό. Όταν εγκρίνει κάποια ιδέα το Κοινοβούλιο και υποστηρίζει ότι θα κινηθεί του το τρόπος για τον προπολογισμό του 2018 και δεν το υλοποιεί εγκρίνουμε κάποια πράγματα που δεν υλοποιούνται μετά. Αυτό είναι απογοητευτικό. Παίρνουμε μια απόφαση, μετά η απόφαση δεν εκτελείται. Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να τονίσω. Πώ να υλοποιούνται οι αποφάσει, εφαρμόζονται οι αποφάσει που παίρνουμε. Μετά μιλήσαμε για, για τα γραφεία ενημέρωση, διάφορε υπηρεσίε του Κοινοβουλίου αναφερθήκαμε στα κέντρα που έχουμε στο Παρίσι, στη Ρώμη κλπ. Και εκεί πρέπει να έχουμε ένα παρλαμεντάριο με ένα γραφείο μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι σταθερό, να υπάρχει ένα κέντρο σταθερό ε, ενημέρωση, να μπορούν να έρχονται επισκέπτε για να μαθαίνουν για την Ευρώπη. Στι μικρέ χώρε θα ήταν μια καλή ιδέα να έχουμε κινητά τέτοια κέντρα του Κοινοβουλίου Παρλαμεντάριου που θα μένουν δύο εβδομάδε, παραδείγματο χάρη για να προσελκύσει παραδείγματος χάρη τους μαθητές, φοιτητές που μπορούν να πάνε και να μαζέψουν πληροφορίες για την Ευρώπη. Και το κινητό μετά παρλαμεντάριο μπορεί να πηγαίνει σε άλλη χώρα. Πρέπει να αναλύσουμε αυτήν την ιδέα, να δούμε πόσο θα κόστιζε ε, μια τέτοια κινητή υπηρεσία ενημέρωση. Ίσως θα μπορούσαμε να το αναλύσουμε και αυτό, αυτό το ενδεχόμενο. Και κάτι άλλο. Ήμουν σκιώδης συζητητής για τον προπολογισμό. Έπρεπε να εγκαταλείψω το καθήκον όμως αυτό. Να σας πω γιατί. Είχαμε παρενόχληση. Είχαμε υποθέσεις ε, παρενόχλησης που εξετάσαμε στο, αντιμετωπίσαμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Είχαμε δεκάδες τέτοιε τέτοιες περιπτώσεις. Ε, εμείς μπορούμε να διαπράττουμε και σφάλματα. Αν δεν γίνονται έρευνες που γίνονται από εμπειρογνώμονες ούτω ώστε να ξέρουμε ακριβώ τι συνέβη, πώ πήγαν τα πράγματα. Αν δεν υπάρχουν εμπειρογνώμονε, μπορεί να διαπράττουμε και σφάλματα. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε αυτού του είδου ειδικού για τέτοιε περιπτώσει. Συζητούμε το έγγραφο, θα συζητήσουμε και το έγγραφο αυτό για την παρενόχληση και θα συζητήσουμε και τα μέτρα τα μελλοντικά στην ομάδα εργασία. Χρειαζόμαστε όμως επαγγελματίες του τομέα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ε, έχουμε ένα, χρειαζόμα, υπάρχει διαμεσολαβητής. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν έρευνες, όπως έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε τέτοιες ε, περιπτώσεις. Ακούνε τους μάρτυρες, χρειάζονται πυρογνώμονες για την εντόπιση των περιπτώσεων παρενόχλησης. δεν μπορούν. Από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο είχα τρει τριμερεί διαλόγου εγώ. Έπρεπε να ακούσω πολλέ μαρτυρίε για αυτέ τι περιπτώσει των παρενοχλήσεων, του harassment. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο ο φόρτο. Γι' αυτό αναγκάστηκα να παραιτηθώ από τη θέση του ηγητού. Σε προηγούμενη θητεία είχαμε περίπου 123 τριμερεί διαλόγου ότι ήμουν ξανά σκιώδη του προπολογισμό. Χρειάζεται να έχουμε εμπειρογνώμονε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό θέλω να πω. Δεν μπορούμε να εργαστούμε που δεν είναι επαγγελματικός. Στον τομέα της παρενόχλησης, του harassment. Με άλλη παρατήρηση. Και στο Προεδρείο συζητήσαμε το θέμα των Αγγλικών. Εγώ δεν είμαι ότι οι Βρετανοί θα φύγουν. Το είπα από την αρχή. Δύσκολη κατάσταση. Ετοιμάζονται. Δεύτερον, θα παραμείνουν για πάντα τα αγγλικά. Επάπειρον θα υπάρχουν τα αγγλικά και να φύγουν οι Άγγλοι. θα είμαστε αφελείς αν πιστεύουμε ότι θα σταματήσει η χρήση των αγγλικών και θα εξαλειφθούν τα αγγλικά. Θα παραμείνουν τα αγγλικά επάπειρον. Αυτό θα πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Μοχόλμαϊρ. Πρόεδρε. Έχω να πω δύο λόγια για την συζήτηση που είχα με τους αρμόδιους. Μπορεί να μην είμαι αρμόδια για τα θέματα της κτηριακής πολιτικής, η οποία έχει τόσο πολύ ταράξει τα νερά, αλλά νομίζω ότι θα ήταν καλό να σε θέση να μπορούμε να προγραμματίζουμε εγκαίρως στον προϋπολογισμό μας και να προβλέπουμε τις ανάγκες. Νομίζω και ο πρόεδρος αυτό προτιμά και θα προσπαθήσουμε κι εμείς να το να ικανοποιήσουμε αυτή την προτίμηση. Όσον αφορά τους ε, ασκουμένους, Μπορεί να έχουμε έναν ασκούμενο από τη συνάδελφη, ο οποίο μπορεί να έρχεται για τρει-τέσσερι εβδομάδες, να χρειάζεται κάποια υποστήριξη ε, για να κάνει τη δουλειά που θα του αναθέσουμε, να χρειάζεται κάποιον βοηθό δίπλα του γιατί είναι για πολύ λίγο καιρό εδώ είναι κάτι διαφορετικό όμως από εκείνον τον ασκούμενο στον οποίο θα δώσουμε μια θέση για ένα, ένα μισή χρόνο και ο οποίος πραγματικά προσφέρει δουλειά βοηθού. Εκεί είναι διαφορετικές συνθήκες και εκεί πρέπει να συζητήσουμε τις δυνατότητες διαφορετικής χρηματοδότησης. Υπάρχουν διαφορετικοί ασκούμενοι που έχουμε συναντήσει και υπάρχουν κάποιοι και είναι εξαιρέσεις βεβαίως που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, που έχουν και νομική κατάρτιση επί παραδείγματι και ε, για τους οποίους καταβάλλεται επειδή είναι σε ένα είδος απόσπασης από τις χώρες τους ο σχετικός μισθός. Είχα εγώ μια τέτοια περίπτωση με 1500 ευρώ ε, μισθό στη Γερμανία και εδώ έπαιρνε μια κάποια, ένα κάποιο συμπληρώμα ε, για έξοδα αλλά πρέπει να προσέχουμε ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτών και των άλλων των ασκουμένων που μπορεί να έχουν μια θέση για ένα-δύο χρόνια και να παίρνουν μια ε, ελάχιστη αποζημίωση, οπότε θα πρέπει βέβαια να προσέξουμε και αυτή τη διάσταση αν τα βγάζουν πέρα. Ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω να στεί κανείς άλλο το λόγο. Νομίζω ότι η ασκούμενη είναι ένα θέμα που θα πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινιστεί. Και βέβαια σε διάκριση μεταξύ εκείνων που ε, πρέπει για ένα-δύο μήνες να κάνουν μια πρακτική εξάσκηση σε ένα από τα θεσμικά όργανα για να ολοκληρώσουν τις σπουδέ τους, οπότε δεν είναι πραγματικοί ασκουμένοι. Κατά κάποιο τρόπο τους καλύπτουμε τα έξοδα διαμονής και από την άλλη υπάρχουν και εκείνοι οι ασκούμενοι οι οποίοι γίνονται, ε, ε, ε υπηρετούν ως βοηθοί των βουλευτών λίγο πολύ. Αλλά το θέμα είναι χρειάζεται ρύθμιση ή πως είναι ένα ζήτημα δεοντολογίας για τον καθένα από εμά. Πρέπει για κάθε τι να ορίζουμε κανόνες και μετά να παραπονιόμαστε ότι είναι περίπλοκα γραφειοκρατικά τα συστήματα, ότι όλο και πεστρούς κανόνες εισάγουμε κτλ. Δεν πρέπει να είναι θέμα δεοντολογίας και να εξαρτάται από την ε, ε, ηθική αξιολόγηση και την δεοντολογία του κάθε βουλευτή το πόσο θα δίνει στον κάθε βοηθό ή ασκούμενο βοήθω. Αλλιώ με, τόσοι, με τόσους κανόνες περιπλέκουν πολύ τα πράγματα. Τριμερεί διάλογοι μα είπε ο κύριο Μάνκα ότι όλο και περισσότεροι γίνονται. Το είπε και ο κύριο Ρουμπίχη, αλλά έχουν τη δική του γραμματεία. Με πολλή δουλειά για του τριμερούς διαλόγους. Υπερβολική θα έλεγα. υπερβολικέ απαιτήσει, άρα πρέπει να κοιτάξετε και τι διοικητικέ ομάδες των διαφορών επιτροπών που ασχολούνται με τέτοια θέματα, κύριε Ισηγητά. Είναι όλο και πιο περίπλοκα τα πράγματα. Είναι πιο εύκολο να κοιτάξουμε τα των βοηθών μας, γιατί ε, είναι η δουλειά τους ξεκάθαρη. Ε, αλλά μην ξεχνάμε και την ε, δουλειά των ε, γραμματιών των επιτροπών. Όλο και περισσότερε κοινέ συνεδριάσει, όλο και περισσότερε συνεδριάσει, απλά και μόνο. Οι τριμερεί διάλογοι και οι ομάδε των επιτροπών μα, και εγώ το βλέπω από τη σκοπιά τη Επιτροπή των Προπολογισμών, σαφώ αυτό, ότι πολύ δύσκολα μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τόση επιβάρυνση. Το 3,9 ναι, μπορούμε να το δικαιολογήσουμε, είναι πιστικό, όπως άλλωστε μας εξήγησε και ο κύριο Ρουμπίχ αλλά ενώπιση των ευρωεκλογών ετοιμαστείτε. Θα το βρείτε μπροστά σας. Γιατί αυτοί που δεν υποστηρίζουν την Ευρώπη, ασφαλώς, θα το αξιοποιήσουν και θα Μπορούσαμε να κάνουμε μια σειρά από εκστρατείες ενημέρωσης και τα λοιπά, ευαισθητοποίησης, αλλά ε, ξέρουμε τι θα επικρατήσει στο δημόσιο διάλογο. Λίγο να το μειώναμε, να το πηγαίναμε στο 3,8. Τέλος πάντων, θα παρακαλέσω τον Παουλ Ρούμπιχ να μας ε, διατυπώσει τα συμπεράγματα για να το ολοκληρώσουμε αυτό και μετά θα πάμε στο επόμενο κομμάτι που θα είναι κυκλισμένο των θυρών και επιτρέψτε μου να αναλάβω να μεταφέρω με τη βοήθεια βέβαια και του κυρίου Μάνκα στο Προεδρείο τη ε, μιλήματά σας ε, για τα έγγραφα διότι να συζητούμε και να λαμβάνουμε αποφάσεις χωρίς έγγραφα δεν γίνεται. Απευθύνω λοιπόν επιστολή στον Πρόεδρο αλλά και το Γενικό Γραμματέα για το θέμα αυτό. Ο δε κύριος Βίλαντ, ο οποίος είναι αναπληρωτής της Επιτροπής μας, θα μας υποστηρίξει, ελπίζω, μαζί με τον κύριο Σασόλη ασφαλώ, ο κύριος Σουριμπή. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους, αλλά και τη γραμματεία για την υποστήριξη. Διότι για μας φυσικά η συζήτηση για τον προπολογισμό του επομένου έτους θα γίνει σε πολύ μεγάλο βάθος και είμαι στη διάθεση όλων σας και για διμερείς επαφές χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτό. Εγώ σας έδωσα μια γενική επισκόπηση τώρα, γιατί ο προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπαίνει σε πολύ μεγάλες λεπτομέρειες και ρυθμίζει πολλά τέτοια θέματα. Γι' αυτό τα όσα είπαν οι συνάδελφοι είναι πολύ σημαντικά για μας και παρακαλώ και στις τροπολογίες να τα διατυπώσετε έτσι ώστε να αναφέρονται τα προβλήματα τα οποία έχουμε εντοπίσει και ε, διαπιστώσει. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε μπει σε αυτή την πορεία και μπορούμε να ρίσουμε και προθεσμοί για την κατάθεση τροπολογιών. Βέβαια, είναι μεγάλη διαφορά αν είσαι από μεγάλη χώρα ή από μικρή. Στη μεγάλη χώρα είναι πολύ ισοπληθισμός και στη μικρή λιγότερος. Το βλέπω εγώ από το δικό μου παράδειγμα, είμαι αρμόδιος για τέσσερις επιτροπές. Και οι δικοί μου βοηθοί φέρουν όλο το βάρος των τεσσάρων επιτροπών. Είπατε και εσείς, Πρόεδρε, ότι οι γραμματείες επίσης είναι επιβαρημένες. Ε, παρόλο που έχουν πάρα πολύ ειδικευμένο προσωπικό, είναι στενά τα περιθώρια. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά ε, για τους υπαλλήλους που έχουμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους μου τους ε, βοηθούς ε, και τους ασκουμένους αλλά και τους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου. Αν μου επιτρέπετε μια μικρή διακοπή, λέει ο Πρόεδρος. Μήπως έχουμε υπερβολικά μεγάλο αριθμό επιτροπών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Äh, Έχουμε 20 επιτροπές τακτικές και αν ε, είναι ο βουλευτής από μια χώρα που έχει 5-6 βουλευτές, τότε θα πρέπει να παρακολουθεί όλα αυτά τα θέματα σε όλες τις επιτροπές και να εξειδικεύεται και σε αυτά και άμα παρακολουθείς τέσσερις επιτροπές είναι σχεδόν αδύνατο να ε, τα παρακολουθείς όλα αυτά σε λεπτομέρειες. Εν πάση περιπτώσει, έλεγα ότι θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με βοήθησαν. Νομίζω ήταν καλή η δουλειά μας και οι αποφάσεις ε, συνενετικές οι περισσότερες σε καλή βάση και με μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Σίγητα. Ε, θα τελειώσει εδώ το ε, δημόσιο σκέλος της συνεδρίασης. Θα διακόψουμε για λίγο και θα προχωρήσουμε σε κεκλεισμένο των θυρών μετά από τρία λεπτά.